Καλημέρα στην ε, πολυάριθμη επιτροπή μας. Έχουμε κοινή συνεδρίαση ΦΑΜ και DEVE σήμερα το πρωί. Και έχουμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο κατάλογο ψηφοφοριών. Να ευχηθώ ένθερμη καλημέρα στον κύριο Τομπέ. Και έχουμε την ε, τιμή να συμπροεδρεύσουμε για μια ακόμη φορά εν ώψη αυτής της νέας ε, νομοθετικής περίοδου θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. So sorry to push now a little bit, but we, we have a long list uh, and I know... Με συγχωρείτε που σας πιέζω, έχουμε μακρύ κατάλογο και ξέρω ότι Πιέζει ο χρόνος ε, και τους συναδέλφους. Καλωσορίζω λοιπόν τα μέλη της ΦΑΜ και της ΤΕΒΕ. Καλημέρα σας ε, και καλή χρονιά σε όσους δεν έχω συναντήσει ακόμη. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλή η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας και είναι πολύ καλό σημείο αφετηρίας ε, Ας ε, περάσουμε και στις ψηφοφορίες και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρέγνερ γιατί έχουμε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Τα βλέπετε και στα αποτελέσματα και ελπίζω να δώσουμε και ένα ισχυρό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τα λόγια αυτά, ας περάσουμε στην ημερησία διάταξη και θα περάσω στα γερμανικά. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά σα. Έγκριση τη ημερήσια ε, διάταξη, όσο δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή να γίνει. Also, <laughs> Να περάσουμε στο 2 της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, αν δεν υπάρχουν ε, αλλαγές, θεωρείται εγκεκριμένη η ημερήσια διάταξη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ένταση. Ελπίζω να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα τώρα. Μάλιστα. Ακούω ότι δεν χρειάζεται να σας ε, ανακοινώσω τις ανακοινώσεις της Προέδρου, γιατί τα διαβάζουν και τα μέλη τη Επιτροπή ΔΕΒ. Δεν χρειάζεται λοιπόν. Και άρα γλιτώνουμε χρόνο. Και έτσι λοιπόν μετά τι ψηφοφορίε θα κάνουν τι ανακοινώσει στα μέλη τη Επιτροπή ε, ΦΑΜ. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να περάσουμε παρά αυτά στι ε, ψηφοφορίε. Μαζί με την ε, Επιτροπή ΜΑΔΕΒΕ, η 25η επέτειο τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη στο διάσκεψη του Νερόμπι ε, καταρχάς σχέδιο προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε λοιπόν. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν ε, ε, είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Παράγραφος 1. Παράγραφος 1 ψηφοφορία κατά τμήματα, την οποία την έχει ζητήσει η ομάδα του ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα. Όλη η παράγραφος χωρίς Sexual and Reproductive Health and Rights. Η κοινή αποστολή λοιπόν για τους ΔΕΒΕ. Έχετε όλα τα στοιχεία μπροστά σας. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Και εδώ ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα από το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παραγράφος 5 πάρει ψηφοφορία κατά τμήματα. Πάλι ζητήθηκε από την ομάδα του ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν έτσι στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Μία ψήφος υπολείπατε. Αν ψήφισατε όλοι σας λοιπόν τώρα. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίνεται. Σχέδιο προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι στην παράγραφο 1, παράγραφος 1, μετά από έτοιμα της του ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. 4. Και πάλι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και εδώ, για την τελευταία τελική ψηφοφορία, θα κάνουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ. Πέρασε. Και πάλι με συντροπτική πλειοψηφία εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στο σχέδιο α, ψηφίσματος. Παράγραφος 1. Η 88 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 9. Για την παράγραφο 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 10 τώρα. Υπέρ. Η συμβαστική 10 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 101. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογία 127. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 106. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται η 108 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται Παραγράφος 4 σε τμήματα ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ υπέρ κατά άποχες Εγκρίνεται. 109. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Να περιμένουμε λίγο ακόμα. Τώρα ψήφισατε όλοι σας. Πέρα ψηφοφορίας λοιπόν. Έγκρινεται. Και περνάμε τώρα στην 110. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 111. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112, 113 και 114. Ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Μας λείπει ακόμα μία ψήφος. Πέρα ψηφοφορίας. 20 είναι υπέρ, 16 κατά εγκρίνεται. 18 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Μάλλον είμαστε πλειοψηφία, αλλά να το ελέγξουμε παρακαλώ. Την 118 παρακαλώ, την ε, επιβεβαιώνουμε, την επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρα ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132. Καταπίπτει. Η επόμενη αυτή. Απορρίφθηκε, συγγνώμη. Άρα, η 132. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 133. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 135 και 138 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 137. Έναξη ψηφοφορίας. 23 ψηφί υπέρ, 20 κατά, εκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην παράγραφο 9. Α, συγγνώμη. Έχουμε πάει παρακάτω. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά γιατί δεν είμαι σίγουρη. Την 139 παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη. Πέρας. 34 κατά, 9 κατά. Ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, αλλά δεν είδα τα χέρια σας παρακαλώ, έτσι πως τα σηκώνονται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 142. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στη συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 192. Υπέρ. Κατά. 192, ναι. Στη σελίδα 9. Υπέρ. 192. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 και 170 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Κάποιες σελίδες παραπέρα στη σελίδα 13. Υπέρ. Για τον συμβιβασμό υπερθμό 13. 15, συγγνώμη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 18. Παράγραφος 18 με χωριστή ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚΑ. Υπέρ. Παράγραφος 18. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186. Υπέρ. Κατά. Ναι, συγγνώμη. Η 186. Άλλη μια φορά. Παρακαλώ να προετοιμάσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172, 189, 190. Από κοινού, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 191. ενενήντα ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 και 194 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο κατάλογος ψηφοφορίας έχει πολύ ακόμα. Ναι, θέλω να σας... Είστε υπομονωτικοί. 197. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 200. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται η 201 α, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη η 202 παρακαλώ λέει η πρόεδρος όχι εγκρίνεται η 202 παρακαλώ υπέρ για τη 202 κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 167 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις αντιλογικές σκέψεις. Recitals. 16. Αντιλογική σκέψη α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 με σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Για την 20. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 και 22 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και έτσι περνάμε στην 27. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην 30 να περάσουμε λοιπόν τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Στις ιδεολογικές σκέψεις πάντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τριάντα επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τριάντα οκτώ. Τροπολογία τριάντα οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία επαριθμών 38 στην αιτιολογική σκέψη FA. Μας λείπει μία ψήφος. 15 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. Και να περάσουμε στην συμβαστική 3, αιτιολογική σκέψη G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, δεν θα ψηφίσουμε το 49, αλλά πάμε στη συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Αντιλογική σκέψη IA. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική έξι. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Επόμενη είναι η τροπολογία 65. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 73. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη π. Ρόλινγκο. Καταπίπτει. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρο. Και φτάνουμε στην ετολογική σκέψη R. 77. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 78. Ο κ. Τραμπέλα, κάτι διαδικαστικό. Για ποιο λόγο καταπίπτει συνέχεια καθώς ε, ε, έχει απορριφθεί η 76 γιατί λέει καταπίπτει ε, αν υιοθετηθεί η 76 ενώ απορρίφθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε για τα δύο μέρη του κειμένου κατά την απόψή μου. Ναι και εγώ αυτό έλεγα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Τραμπέλα. Να ψηφίσουμε λοιπόν την εκλογική σκέψη π. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. σα ευχαριστώ πάρα πολύ. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο S79. Τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τάφε 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιου τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβαστική 8 Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, διορθώνει η πρόεδρος. Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην 85. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στα citation. 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Βλέπω ότι είναι ταυτόσιμη με τη 2. τροπολογία υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες να ελέγξουμε. Έναρξη. Παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Στην τροπολογία 3, στις αυτολογικές αναφορές. Πέρα ψηφορία. 25 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική 1. Στι λογικέ αναφορέ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. 12 και 13. Ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Με τα χέρια σας Υπέρ παρακαλώ της 8. Ε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14. Α, συγγνώμη λέει, πρόεδρος, συγγνώμη. Εγκρίθηκε η συμβαστική παραθμών 2 και έτσι μετά από μια μακρά ψηφοφορία να περάσουμε και στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας και όπως βλέπετε 39 είναι οι ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά, 3 οι αποχές. Να, μας συγχαρούμε, να σας συγχαρώ όλους σας, να σας συγχαρώ για την ενεργή συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ψηφοφορία. Και να ευχαριστήσω και τους συναδελφούς της Επιτροπής Ανάπτυξης για τη συμμετοχή τους. Και θα ήθελα και εγώ να πω προς όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ΔΕΒΕ, σας παρακαλώ βγείτε γρήγορα από την αίθουσα. So it was not on the micro we realized. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά καταλάβατε καλά. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της ΔΕΒΕ και όλοι καλούνται να πάνε στις ε, αντίστοιχες συνεδριάσεις τους. Διακόπτουμε τη δική μας Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών για ένα δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τόμπε. So, uh, Κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι κάθονται ήδη τα μέλη και περιμένουν να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες. Είμαστε στη μέση των ψηφοφοριών. Σας, ζητώ παρακαλώ να καθίσετε και να διακόψετε τις συζητήσεις για να μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Και να μιλήσω πάλι γερμανικά. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή. 2018 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. EIGE. E. Ψηφίζουμε λοιπόν και να ξεκινήσουμε με την συμβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος. Συμβαστική 2 μάλλον. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 9 παρακαλώ. Ψηφίζουμε την τροπολογία αριθμό 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4α. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Τη Βιλία Μπλίκεβιτσιούτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία υπερθμών 20. Πέρας. 15 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται τα 20. λογική σκέψεις. Β. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά, όπως πάντα, έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μόνο 25 ψηφίζουν. 20 υπέρ, 5 κατά. Συγχαρητήρια. Και συνεχίζουμε με την απαλλαγή. 2018, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ να ξεκινήσουμε με τη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτάκι. Συμβαστική τρία τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τέσσερα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αντιλογικές ε, σκέψεις ε. συμβαστική 5 καταρχάς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και εδώ η τελική ψηφοφορία, παρακαλώ, ηλεκτρονικά έναρξη. Πέρας, 19 υπέρ, 5 κατά, συγχαρητήρια. Και εδώ ολοκληρώθηκε και αυτό το κεφάλαιο με επιτυχία. Και περνάμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, απασχόληση και κοινωνικέ πτυχέ στην ετήσια επισκόπηση τη ανάπτυξη για το 2020. Και ξεκινάμε την ψηφοφορία μα. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν ε, κατάλαβα το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το ξανακοιτάξουμε. Να ελέγξουμε παρακαλώ λοιπόν την 18. Λείπει μία ψήφος. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν, ναι. Η 20 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 29. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέραψη φορέας, 14 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η 33. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλά την 41. Ε, Περάς. 15 υπέρ, 9 κατά. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές με την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 45 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά το ελέγξουμε παρακαλώ. Τη 45 παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν έχει κλείσει ακόμα η ψηφοφορία. Μα τι γίνεται, όλο και πιο λίγοι συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. 10 υπέρ, 12 κατά. Απορρίπτεται. Η 46 υπέρ. Κατά. Η ίδια ισορροπία απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Η 52. Τροπολογία 52, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 52. 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 12 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, ας ελέγξουμε παρακαλώ. Την 60 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τώρα κάπως παραπάνω ψήφισαν. Πέρα ψηφορία. 19 υπέρ, 5 κατά. Σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 64. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Πέρασε τώρα. 10 υπέρ, 12 κατά, απορρίπτεται. 65 λοιπόν τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις θετολογικές σκέψεις. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τροπολογία 8. Ρόζα Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Με σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Για την 13 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, δεν περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία αλλά ολοκληρώνεται η ψηφοφορία αυτή. Και εδώ να συγχαρώ την κυρία Καλβές. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ όμως για την επιμονή σας και την υπομονή σας. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε μία ακόμη. Προφορική ερώτηση για τις προτεραιότητες ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την 64η Σύνοδο τη Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση τη γυναίκα. Και να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας. Παράγραφος 2. Πρώτη παύλα. Μία τροπολογία του ID. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Τρίτη. Παύλα. Του ECR παρακαλώ πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. ΕΛΚ, ECR και ID. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο τρίτο τμήμα. Από το ID πάλι. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Παράγραφος 3. ID. Η διαγραφή των λέξεων following the priorities και το καθεξής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Και τώρα στην παράγραφο 4. Τεχνική. Τροπολογία. Υπέρ. Α, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε αυτή, μια σκηνή τεχνική τροπολογία. Δεν προβλέπεται ψήφιση. Τελειώσαμε λοιπόν με τις τροπολογίες να κάνουμε την τελική ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορίας. 18 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, Εγκρίνεται η προφορική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ πειταρχημένη ψηφοφορία. Πέρας των ψηφοφοριών. So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σημεία στην ημερησία διάταξη. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που έχουμε ως προσκεκλημένη την Υπουργό Δημογραφίας, Οικογένειας και Νεολαίας της Κροατίας, την κυρία Βέσνα Μπεντέκοβιτς θα ήθελα και πάλι να σας ε, ζητήσω να φορέσετε τα ακουστικά σας, γιατί θα μιλήσω γερμανικά. So, also, äh, sehr geehrte Mitglieder, wir gehen jetzt... Äh, Αγαπητοί βουλευτές, να συνεχίσουμε μετά τις ψηφοφορίες. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Βέσνα Πεντέκοβιτς, ε, Υπουργό της Κροατίας για Δημογραφία, Οικογένεια και Νεολαία. Η Κροατική Προεδρία ανυπομονούσαμε να ακούσουμε το πρόγραμμά της για τα θέματα ισότητας και πολλές είναι οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα είναι πραγματικά συναρπαστική η κυρία μα, Πρωτού δώσω το λόγο στην ε, Υπουργό να κάνω κάποιε παρατηρήσει ε, οργανωτικής φύσεως, ε. μιας και είχαμε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της επιτροπή ΔΕΒΕ, δεν σα έκανα τι ανακοινώσει που αναλογούσαν στην Επιτροπή ΦΕΜ. Θα τι ακούσουμε λοιπόν τι ανακοινώσει μετά την παρουσίαση της Υπουργού της Κροατίας. Λίγο λοιπόν πριν από το τέλος θα σας ε, διαβάσω και τις ανακοινώσεις για την Επιτροπή μας. Τώρα, για την Κροατική Προεδρία, ανυπομονούμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η υπουργό. Θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Κροατικής Προεδρίας η υπουργό. Μετά θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους ε, των πολιτικών ομάδων και προφανώς σε όλους τους υπόλοιπους και μετά από τις ερωτήσεις αυτές θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Σας καλωσορίζω εκ νέου στην Επιτροπή μας και έχετε το λόγο. So much now. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να συνεχίσω στα κρατικά. Αξιότιμη πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμοι συντονιστές των πολιτικών ομάδων, μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ότι καταρχάς είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω ως εκπρόσωπος της κρατικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τα γνωρίζετε, η Κροατία μετά από 6,5 χρόνια συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο φρέσκια χώρα που έχει αναλάβει τα ενία της Προεδρίας και αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας. Και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία και τους τομείς δραστηριότητας της κρατικής προεδρίας σε ό,τι αφορά το θέμα της ισότητας των φύλων. Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας βασίζεται στις κοινέ ευρωπαϊκές ε, αξίες και το σεβασμό των ε, κοινών μας συμφερόντων. Στο επίκεντρο του προγραμματός μας είναι ο πολίτης. Οι ανάγκες, οι προσδοκίες του πολίτη, η ασφάλεια και το βιωτικό επίπεδο, η ποιότητα ζωής του πολίτη. Θα να σκέψουμε λοιπόν στους τομείς αυτούς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία και παράλληλα θέλουμε να τονώσουμε το αίσθημα του αλληλοσεβασμού και του σεβασμού των κοινών αξιών. Τους πρώτους λοιπόν έξι μήνες του τρέχοντος έτους θα εργαστούμε πυρετοδός για να προωθήσουμε αυτή την ισχυρή Ευρώπη. Και γι' αυτό λοιπόν η εξάμενη προεδρία μας θα ακολουθήσει το συνθήμα μια ισχυρή Ευρώπη σε μια και μια ενωμένη Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν τις ε, προτεραιότητες ε, για μια Ευρώπη η οποία ενώνει, που προστατεύει, που ενισχύει και που έχει επιρροή. Σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκείται για την ισότητα των δύο φύλων και την ε, ίση συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Θα θέλαμε να προωθήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία και θα θέλαμε να ενισχύσουμε την ανεξαρτή απασχόληση των γυναικών, γιατί αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και κυρίω θα ασχοληθούμε με θέματα συνοχή. και να δούμε τι σύνδεση υπάρχει με τη μη ασχολησιμότητα κάποιων γυναικών και με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αυτέ οι γυναίκε για τη συμμετοχή του στην αγορά εργασία. Θα ανελύσουμε λοιπόν τι προκλήσει αυτέ και θα προτείνουμε σχετικέ λύσει. για να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των γυναικών και προκειμένου να μπορέσουν να συμμετέχουν επίση όρες στην αγορά εργασία. Θα προσπαθήσουμε όλους ιδιαίτερω να εξακριβώσουμε και το πρόβλημα τη γύρανση του πληθυσμού πώς διαμορφώνεται, καθώς ε, και της ε, μακροχρόνιας φροντίδας ε, μελών της οικογένειας και πώς συνδέεται πάλι αυτό με την χαμηλή απασχολησιμότητα των γυναικών. Θα καταθέσουμε λοιπόν σχετικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής και της δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, εδώ θα προσπαθήσουμε να βρούμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου και θα διοργανώσουμε και διάφορε εκδηλώσει για την προώθηση των προτεραιοτήτων μα. Θα κάνουμε τέλη Ιανουαρίου, για παράδειγμα, μια διάσκεψη για το θέμα τη υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Συμμετοχή λοιπόν των γυναικών στην αγορά εργασία, όφελο για όλη την κοινωνία. Αυτό θα, αυτός θα είναι ο τίτλο και θα θέλαμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να απαλείψουμε τα εμπόδια που στέκονται στο δρόμο των γυναικών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί. Οι προκλήσεις λοιπόν με τις οποίες ε, θα ασχοληθούμε είναι οι εξή. Πώς μπορούμε η ανάγκη και η ζήτηση στην αγορά εργασίας να έχουν καλύτερη αντιστοίχηση, βιωτικό, επαγγελματικό και οικογενειακό βίο, σεξουαλική παρενόχληση στην αγορά εργασία, μακροχρόνια φροντίδα των ε, μέλων τη οικογένεια και στη διάσκεψη λοιπόν θα συμμετέχουν ε, μέλη από τα κράτη-μέλη, από την κοινωνία των πολιτών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλη των ακαδημαϊκών κύκλων. Έχουμε λοιπόν και τα απορίσματα του Συμβουλίου, τα οποία θα πρέπει να, τα οποία θα πρέπει να καταρτήσουμε για τη μακροπρόθεσμη λοιπόν φροντίδα και το πώς επηρεάζει την ε, σύνδεση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Με σκοπό φυσικά να έχουν τελικά ίση συμμετοχή οι γυναίκες ε, στην αγορά εργασία. προκειμένου αυτή η μακροπρόθεσμη φροντίδα να είναι κάτι το εφικτό για όλους θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τους πολιτικούς μας στόχους για να δούμε πώς μπορούν να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές στην κοινωνία και πώς μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή, ένας σοβαρής καταμερισμός των ευθυνών αυτών. Θα θέλαμε επίσης να ενημερώνουμε και να ενημερώσουμε καλύτερα τους πολίτες για τα ήδη φυστάμενα μέσα και μέτρα για την καλύτερη υποστήριξη επαγγελματικού και οικονομικού και οικογενειακού βίου. Επίση, στη διάσκεψη αυτή για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία θα συζητήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα υποβάλουμε και μία μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Αυτό θα αποτελέσει και τη βάση των πορισμάτων. Και στο επίκεντρο φυσικά θα είναι η ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει βασικό στόχο τη κρατική προεδρία για τα θέματα ισότητα των φύλων και θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι δεν θα περιοριστούν οι προσπάθειέ μα ε, στο σημείο αυτό και στη διάσκεψη αυτή. Έχουμε περαιτέρω προκλήσει ε, για το μέλλον και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι, όλοι να αγωνιστούν για την ε, εξασφάλιση και προώθηση και ενίσχυση τη ισότητα των φύλων. Όχι μόνο δηλαδή η κρατική προεδρία, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί, όλοι οι παραγόντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συμβάλλουν προ την κατεύθυνση αυτή. Η κοινωνία των πολιτών, τα θεσμικά όργανα, είμαστε όλοι εταίροι στην προσπάθεια αυτή. Είμαστε λοιπόν στην αρχή μια νέα θεσμική περίοδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα πολιτική βούληση και αυτό αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης για τις περαιτέρω βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να γίνει α, αυτό το gender mainstreaming. Η εγκάρσια δηλαδή προάσπιση τη ισότητα των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανδρών σε όλες τις πολιτικές. Θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση για όλου σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε συνέχεια, ε, συνοχή και επιμονή. Και νομίζω ότι μόνο αν ε, δράσουμε βάσει ενό σχεδίου δεδομένων και των νέων προκλήσεων, των νέων συνθήκων, αν ε, αναζητήσουμε τι ε, βαθύτερε αιτίε τη ανισότητα μεταξύ των φύλων, θα μπορέσουμε τελικά να σχηματίσουμε μια κοινωνία πιο ίση. Αλλάζει ταχαίως ο κόσμο μας και θα πρέπει διαρκώς να αντιλαμβανόμαστε τις ε, προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Και με όλα αυτά λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλό μας θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ουδέτεροι και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να πετύχουμε καλύτερη ευημερία για όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι δεπεπισμένη, όπω άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι φορεί και όλοι οι υπόλοιποι στην Προεδρία, ότι θα είναι εξαιρετική συνεργασία για όλε αυτέ τι μελλοντικέ προκλήσει. Σα ευχαριστώ και όλα αυτά τα είπα εντελώ εισαγωγικά και προσβλέπω φυσικά στις ερωτήσεις από πλευρά σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισαγωγική σας αυτή παρουσίαση σε σχέση με το πρόγραμμα της κρατικής προεδρίας και θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές μας. Από πλευρά του ΕΛΚ, η Ελισαμπέτα Λουκαβιέτσκα. Πείτε. Yes. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για μας τις γυναίκες. Έχω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν, έχοντας κατά νου ότι μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας ε, είναι η καταπολέμηση των δημογραφικών προκλήσεων. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες. Ποια είναι τα σχέδια της Προεδρίας σας για το θέμα αυτό. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η θέση σας ε, για το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι συγκεκριμένες προκλήσεις ε, στην εποχή ε, της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική για την ισότητα και πώς θα βοηθήσετε τις γυναίκες με αναπηρία. Και τέλος, μπορείτε να μας πείτε τι θα συμπεριλαμβάνετε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το συσχετισμό ε, μεταξύ των γυναικών στην αγορά εργασίας ε, και της υποχρέωσης μακρόχρονης μέρημνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλήθος ερωτήσεων. Και να περάσουμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Μάτιτς. Ε, thank you, Evelyn. I will... Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα κρατικά. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σα αυτή και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων τη κρατική προεδρία. Και διάβασα προφανώ τι ε, προκαταρτικέ δηλώσει τη κρατική προεδρία. Μία από τι βασικέ προτεραιότητε είναι το θέμα των δημογραφικών αλλαγών. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η κυρία Σουίτσα είναι και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια για θέματα δημογραφία. Σε ό,τι αφορά τη δημογραφία λοιπόν και τι προτεραιότητε αυτέ, θα θέλατε ίσω να μας εξηγήσετε λίγο πιο αναλυτικά πώς αυτά θα έχουν επιπτώσεις στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και πώς διαμορφώνεται αυτό στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος από την ομάδα του Ρινιού, η κυρία Μαρία Ροντρίγκης Μαραμό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων υπό την Προεδρία σας. Και θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και καλά αποτελέσματα για το επόμενο εξάμεινο. Διάβασα και τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας και σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα, που αποτελεί τη δεύτερη προτεραιότητα. αυτό ο ευρωπαϊκό Πυλώνας είναι ιδιαίτερα ευρύ. και αναφέρεται στην πλήρη ένταξη, στην ισότητα και στη συμμετοχή στην αγορά εργασία ε, και στην πρόοδο στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό το δικαίωμα στην ισότητα δυστυχώς πλήττεται στα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από το ΕΓΚΕ μας λένε ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ίδια θέση, με ίδιες ευθύνε είναι 20% και η διαφορά εσόδων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις συντάξεις που λαμβάνουν είναι της τάξης του 35%. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας έχετε σκεφτεί να προσεγγίσετε κάποιο μέτρο ή να δώσετε κάποια συγκεκριμένη όθηση. Γιατί θα πρέπει ταχύτατα να καλύψουμε αυτό το μισθολογικό χάσμα. Δεν ε, μπορούμε να το κληροδοτήσουμε και στις κόρες μας, ε, γιατί ε, πρόκειται εδώ για παραβίαση του δικαιώματος της ισότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων για λόγους φύλου. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω αν στις προτεραιότητές σας έχετε σκεφτεί να προσεγγίσετε κάτι που είναι θεμελιώδες για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας. Δηλαδή, οι χώρε που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, Λιθουανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Λετωνία, να το κάνουν ταχύτατα. Τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου μα λένε ότι για να καταπολεμήσουμε την έμφυλη είναι απαραίτητο να έχουμε διεθνή μέσα και η σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Καλή τύχη με την Προεδρία σας, γιατί αν έχετε εσείς επιτυχία θα είναι και δική μας. Äh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο στους πράσινους. Η Γκουέντολιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Διαναφέρθηκε η δημογραφική αλλαγή είναι μια νέα προτεραιότητα της Κομισιόν ο τίτλος ε, «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής» προκάλεσε πολλές συζητήσει, αλλά σε ό,τι με αφορά στους Πρεσίνου ε, και μας, μας εξέπληξε ε, ο τίτλος «Δημογραφία και Δημοκρατία». Είναι αρμόδια είναι αρμοδίο ο Κροάτη Επίτροπο για το χαρτοφυλάκιο αυτό. Και βέβαια αυτά τα θέματα επανέρχονται στη συζήτησή μα. Σε κάποια κράτη έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα με τη γύριανση του πληθυσμού και με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Βέβαια, αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και είναι μια συγκεκριμένη ανησυχία που έχουμε. Ξέρουμε ότι θέλετε να οργανώσετε την Άνοιξη μια σύνοδο για τη δημογραφία. Ποια θέματα θα συζητηθούν στη σύνοδο αυτή και τι θα παρουσιάσετε στο θέμα της δημογραφίας. Ε, η δημογραφική ζωτικότητα χρησιμοποιείται πολλές φορές από τον κύριο Όρμπαν π.χ. στην Ουγγαρία κατά της μετανάστευσης. Ε, λέει ότι ε, δεν θέλουν να υποδεχτούν μετανάστες, αλλά θέλουν περισσότερους εθνικούς υπήκους. Θα αναφερθείτε εσείς σε αυτό το θέμα γιατί μας ανησυχεί και επίσης βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται το θέμα της δημογραφίας σε συντηρητικούς πολιτικούς λόγους ε, για να παρουσιάσουν μία λευκή οικογένεια ε, ετεροφιλόφιλη. Έτσι λοιπόν ε, χρησιμοποιούνται αυτά για την πρόθεση της ξενοφοβίας και της ομοφοβίας. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή ήταν η πρώτη ανησυχία που είχα εγώ όταν άκουσα τη συσχέτιση των λέξεων δημοκρατίας και δημογραφίας. Πίσω από αυτή την ε, ανησυχία μπορεί να κρύβεται η επίθεση κατά των αρπαρογικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων για να υπάρχει μια ελεγχόμενη δημοκρατία. Έτσι λοιπόν το θέμα της δημογραφίας χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο των σωμάτων των γυναικών. Ελπίζουμε να μας καθισχάσετε στις σχέση με τα θέματα αυτά. Πολλές ερωτήσει και να δώσω το λόγο από πλευρά της ΓΚΟΕ στην κυρία Ροντρίγκε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ για να μιλήσετε στα μέλη της Επιτροπής μας. Αντίστοιχα με την ε, συνάδελφο από τους Πρασίνους, ε, πρέπει να πω ότι η Κροατία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα δημογραφικά ζητήματα και θα ήθελε το δημογραφικό να ενταχθεί στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μία από τις προτεραιότητές σας. Δεν μας εκπλήσει βεβαίως, ε, διότι υπάρχουν προβλήματα, ιδιαίτερα σε ε, ορισμένες χώρες που είναι χαμηλό το ποσοστό των γεννήσεων και αυτό φυσικά μπορεί να επηρεάσει και τη ζωή και την ε, ε, φορολογική επιβίωση. Και φυσικά αυτό ανησυχεί και κάποια τμήματα στην κοινωνία των πολιτών που λέει ότι υπάρχει και μεγάλη παναχώρηση για σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Μας ανησυχεί ότι προσφάτως στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρο εισήχθησαν θέματα ε, για το δημογραφικό, στο οποίο είναι αρμόδιος ένας καθηγητής, ο οποίος είναι γνωστός ακροδεξιός. Και πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον Ορμπάν και την ε, ε, Ουγγαρία και είχαμε κάποιες θέσεις σε ένα κογκρέσο που έγινε στη Βουδαπέστη τον Οκτώβριο, όπου υπήρχαμε σαφείς πολιτικές διακρίσεων και μάλιστα και αποκλειστικά χριστιανικά. Μια πολιτική λοιπόν η οποία είναι αμυγός ε, ξενοφοβική και ακούστηκε ότι θα μπορούσε να μειωθεί το ποσοστό ε, των μεταναστών και φυσικά αναφέρθηκαν μόνο συμβατικές οικογένειες με πατέρα, μητέρα και παιδιά. Θα θέλαμε να μας καθησυχάσετε εσείς και να μας πείτε ότι όλα αυτά δεν συνάδουν ε, με τη δική σας τη στάση όσον αφορά τα δημογραφικά ζητήματα. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε εσείς το δημογραφικό ζήτημα. Επίσης, ε, θα ήθελα να ξέρω τι μέτρα σκοπεύετε να εφαρμόσετε για να λύσετε τα δημογραφικά προβλήματα, το χαμολό ποσοστό γεννήσεων επίσης ε, και θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να μειώσουμε και τις ανεπιθύμητες ε, να έχουμε πολιτικές γεννητικότητα υπεύθυνε, οι οποίε εγγύονται τα ίδια δικαιώματα σε άνδρες και γυναίκε για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματο. Τέλο, μήπω πιστεύετε ότι οι μετανάστε ε, που έρχονται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μια λύση για αυτό το πρόβλημα τη γύρανση ε, του πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία μελήτρια από το ID, η Άνικα Ρίνερ και μετά θα δώσω το λόγο στην Υπουργό και μετά θα ακούσουμε το δεύτερο γύρο και το λόγο θα έχουν ε, ε, πάλι η Ελισαπέτα και στο τέλος θα κάνω και εγώ μία ερώτηση για να κάνουμε έτσι δύο γύρους ερωτήσεων ιδάλλως τα πράγματα ενδεχομένω να είναι πολύ δύσκολα για την Υπουργό. Άνικα Μπρίνερ λοιπόν τώρα. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Η ερώτηση μου κυρίως αφορά την ε, επαγγελματική βίο, ε, ε, ζωή. Γνωρίζοντας τι συμβαίνει στην Κροασία εδώ και 50 χρόνια, που αφορά και τους άντρες, η ασφάλεια στην εργασία, αμοιβέ οι οποίε δεν δίνονται στην εργασία. Θα ήθελα να ξέρω τι λύσεις ε, ε, σκέφτεστε, διότι υπάρχουν αρκετέ δυσκολίε για να μπορέσουν να ενταχθούν οι γυναίκες ε, στον εργασιακό βίο. Τι μέτρα λοιπόν πρέπει να λάβετε, δεδομένου ότι υπάρχουν και δυσκολίες στην Κροατία και για τους άντρες στο επαγγελματικό περιβάλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. E, Ευχαριστώ πολύ. Για να προσπαθήσουμε να μαθαποίησουμε λίγο τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Να προσπαθήσουμε λοιπόν θεματικά να πραγματευτούμε τα θέματα αυτά. Σημείωσα διάφορες ερωτήσεις και έτσι θα προσπαθήσω με μία απάντηση να δώσω λεπτομέρειες για διάφορες ερωτήσεις. Καταρχάς, μία ομάδα ερωτήσεων αναφορικά με τις δημογραφικές εξελίξεις. Χαίρομαι που κάνατε αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. γιατί οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τις προκλήσεις αναφορικά με την δημογραφική αλλαγή. Και αυτό καταδεικνύει εκ νέου πόσο μεγάλε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνεται εδώ και το γεγονό ότι στη διάρκεια της προεδρίας ε, της Κροατική προεδρίας ε, αποφασίσαμε να καταρτήσουμε τις προτεραιότητές μας ε, και ότι ίσως τα κάναμε και βάλαμε το θέμα αυτό ανάμεσα στις προτεραιότητες μας, γιατί περίπου το ίμιση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη δημογραφική αλλαγή και τις δημογραφικές τάσεις που παρατηρούνται. Μιλώντας λοιπόν ε, για το θέμα αυτό, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, διαπιστώνουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν ε, ακριβώς τα ίδια προβλήματα όλες ε, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι οι ίδιες οι τάσεις πάντα. Κάθε σύσταση λοιπόν και κάθε προφανής ε, λύση στα θέματα αυτά θα πρέπει να εμπεριέχει και την απαραίτητη ευελιξία. Θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο να παρατηρηθούν οι δημογραφικέ ιδιαιτερότητε και να δεχτούν προφανώ υπόψη. Ενώ διαρκώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση και την βελτίωση τη ευρωπαϊκή αυτή ε, διάσταση. εκφράσατε ανησυχία για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των ε, γυναικών, τα δικαιώματα των ε, μεταναστριών, ε, τα θέματα τα οικογενειακά και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις δημογραφικές εξελίξεις. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω αυτές εξ αρχής ότι σήμερα εδώ βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της κρατικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έρχομαι να σας μιλήσω ως ε, αρμόδια υπουργό ε, της Κροατίας για τα ζητήματα αυτά. Το ερώτημα αυτό που θέσατε είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κατανοώ τις ανησυχίες σας και όλα τα σχετικά σημεία τα οποία τα επισημάνετε και εσείς ο ίδιος. Έχουν να κάνουν όμως με το εθνικό συγκείμενο, το οποίο ε, με χαρά μου να το συζητήσω διμερός μαζί σας μετά τη συνεδρίαση, εφόσον έχουμε την ευκαιρία. Σήμερα όμως βρισκόμαι εδώ στην Επιτροπή σας ως εκπρόσωπος εξοχήν της Κροατικής Προεδρίας και όχι ως Υπουργός Εθνική για τα θέματα οικογένειας και νεολαίας της Κροατίας. Τώρα, να δούμε λοιπόν την Κροατική Προεδρία και το θέμα της ε, δημογραφίας, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα. Να τονίσω στο σημείο αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, ότι το θέμα αυτό για πρώτη φορά μπαίνει στη στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αυρία συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές εξελίξεις, σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές πολιτικές. Για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών να έχουμε καλύτερη σχέση με την επαγγελματική ζωή και ούτω καθεξής. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν καταρχάς να κάνουμε μία ανάλυση της κατάστασης και μία περιγραφή της κατάστασης προκειμένου να γίνει μία ευρεία συζήτηση βάσει δεδομένων όμως σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και όλα τα κρατη να μπορέσουν να επισημαίνουν τα τις ανησυχίες τους. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη, τις ανησυχίες τους, τις ιδιαιτερότητές τους. Θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε και βέλτιστες πρακτικές από τα κρατη εφόσον επιθυμούν να μας τις ανακοινώσουν. Γιατί προφανώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που θέλουμε να θέσουμε στο επίκεντρο. Θέλουμε να προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού αυτού να αναλύσουμε τις ε, διάφορες δημογραφικές τάσεις και να απαλύνουμε τις τάσεις εκείνες που μας ανησυχούν προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη όλων των κρατών μελών. Και εδώ προφανώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού σε κάποια κράτη-μέλη. Μιλώντας ε, για τη γύρανση του πληθυσμού και για δημογραφικά τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει να είμαστε άκρος θεωρώ, και να συνειδητοποιήσουμε και να υπενθυμίσουμε στους πολίτες μας ότι όλα τα κρατημέλη πλήττονται από τα φαινόμενα αυτά. Η κρατική προεδρία λοιπόν αντιλαμβάνεται τα ζητήματα αυτά. Γιατί αυτό προφανώς ε, ε, έχει επιδράσεις και στις ε, δημογραφικές εξελίξεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη γύρανση του πληθυσμού. Να επιστρέψουμε τώρα στο επόμενο θέμα, σε ό,τι αφορά το συμβιβασμό της οικογενειακής ζωής και της επαγγελματικής ζωής. Κάντε εδώ πέρα κάποιες ερωτήσεις και πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Βασικό θέμα λοιπόν. Μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία και φυσικά ο σκοπό μα είναι να δημιουργήσουμε καλύτερε συνθήκε για τη συμμετοχή αυτή στην αγορά εργασία. Όχι όμω ό,τι αφορά την συμμετοχή στην αγορά εργασία, αλλά και οι καλύτερε συνθήκε και οι καλύτεροι όροι για την ε, συμφελίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Εδώ θα πρέπει να αναλάβουμε, να αναλάβουμε μέτρα τα οποία θα έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της οικογένειας στην κοινωνία και προφανώς τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κάθε αυτήν όλων των πολιτών μας. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξή. Την αρχή της ισότητας η οποία διαρκώς θα πρέπει να διαφυλάτεται. Και όταν μιλάμε για την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Άλλο ένα θέμα φυσικά σημαντικό είναι το θέμα τη μετανάστευση. Όταν μιλάμε για μετανάστευση στο ευρωπαϊκό χώρο, θα ήθελα να θέσουμε και να κοιτάξουμε ένα επιπλέον θέμα. Δεν είναι τόσο ερώτηση αυτή που θα ήθελα να απευθύνω, αλλά πιο πολύ μια πρόκληση. Το θέμα της κινητικότητας. Των ανθρώπων σε Νέα ηλικίε των νέων, του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυνατότητα λοιπόν μετακίνησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς βασίζεται στην αξία και στην αρχή αυτή της ε, ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών. Και στο πλαίσιο αυτό, μια ενεργή πολιτική μετανάστευσης είναι απολύτως απαραίτητο, απαραίτητη και προφανώς βασίζεται στην αξιοπρέπεια, σε όλες τις αρχές και τις αξίες που είναι σημαντικές για μας. Και σε ό,τι αφορά την πολιτισμική εξέλιξη των κρατών μελών, για το θέμα τη μετανάστευση και το θέμα τη κινητικότητα τη ελεύθερη μετακίνηση στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά επηρεάζει όλες ε, τις πτυχές της ε, ανάπτυξης και προϋποθέτει και μία εγκάρσια ε, διαμόρφωση των πολιτικών. Στο πλαίσιο τώρα της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών, το οποίο αποτελεί και εκτιμένο δικαίωμα προφανώς, έχουμε να επισημάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν για την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί ω τάση, θα πρέπει να το ενισχύσουμε περαιτέρω. Η Κροατία, η Κροατική Προεδρία σίγουρα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο τώρα των δημογραφικών προκλήσεων, Ακούσαμε και μία υπερτερή ερώτηση. Το θέμα που δείξατε κι εσείς για τη βελτίωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γενικών. Προφανώς αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύονται. Δεν χωρά αμφιβολία. Και στο σημείο αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω την προστασία της σεξουαλικής ε, και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων αυτών των γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής και διεθνούς στρατηγικής και εθνικής στρατηγικής. Είναι ύψης της σημασίας να υπάρχει πλήρης προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Ακολουθώντας φυσικά και τις ε, προδιαγραφές που ήδη υφίστανται από την νομοθεσία. Εδώ θα χρειαστεί περαιτέρω ευαισθητοποίηση για όλους τους ε, παραγόντες και φορείς ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθεί, να υπάρξει πρόοδος και στον τομέα αυτό. Τώρα, ασφαλώς και η καθημερινότητα μας αποδεικνύει ότι εδώ θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω τη σύνοδο στο Ναϊρόμπι και την πρωτοβουλία που έθεσε σε, αποτέλεσε την αρχή διαφόρων πρωτοβουλειών σε ό,τι αφορά τη ζωή των γυναικών, στη ζωή των κοριτσιών. Και σε ό,τι αφορά το θέμα του αποκλεισμού εδώ, να υπενθυμίσουμε και θέματα εφαρμογής του προγράμματος τη Διεθνούς διάσκεψη για την Ανάπτυξη και τον Πληθυσμό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του ΟΗΕ. Και εδώ να επισημάνουμε και τους στόχους της βιώσιμη ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τη σύνοδο αυτή. Ένα μεγάλο ζήτημα ήταν το ζήτημα της δημογραφίας. Και στο πλαίσιο αυτό της Συνόδου στο Ναϊρόμπι. Θα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα της, ε, των γυναικών, να συνεχίσουμε τις πρόοδους προς την κατεύθυνση αυτή, για να ξεπεράσουμε και τις δημογραφικές προκλήσεις που έχουν ε, προφανώς επιπτώσεις και στο σκέλος αυτό. Και εκ νέου να τονίσω ότι θα πρέπει να τράσουμε από κοινού. Βέβαια, εδώ θα υπογραμμίσουμε και το δικαίωμα επιλογής κοριτσιών και γυναικών για το πώς θέλουν να ζήσουν. Ακούσαμε άλλη μια ερώτηση σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ήταν δική σας η ερώτηση. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Προφανώ και θα πρέπει να συνδεθεί με τη μελλοντική οικονομική πολιτική. Αυτό αποτελεί μία από τι προτεραιότητε τη ε, Προεδρία μα. Και στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο τη στρατηγική ε, στρατηγικής μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει συνέχεια πρόοδο ενίσχυση. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει αυτή η βιωσιμότητα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια στρατηγική πολιτική, όπω είπα, και να είμαστε συστηματικοί. Με πλήρη δέσμευση να ταχθούμε στο σκοπό αυτό. Και αυτό αφορά όλους τους παράγοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάπτυξη συνεργασιών επίσης μεταξύ οικονομικής και κοινωνική πολιτικής θα πρέπει να υπάρξει. Εδώ λοιπόν υπογραμμίζουμε εκ νέου τις αρχές του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Και πάλι, να είμαστε ρεαλιστές πάνω απ' όλα. Και να αντιληφθούμε ότι παρά τις θετικέ εξελίξεις, ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και ένδιας εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερος δε όταν μιλάμε για παιδιά νέους, ανάπηρους, μέλη εθνικών και λοιπόν μειονοτήτων και προφανώς και μετανάστες. Αυτές οι ομάδες του πληθυσμού αντιμετωπίζουν ιδιαίτερω προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, σε όλους τους άλλους τομείς ε, της κοινωνίας. Και άρα και αυτές οι κατηγορίες των πολιτών θα χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. το θέμα του εισοδήματο προφανώς είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να επέλθει μεγαλύτερη ισορροπία, αλλά αντιμετωπίζουμε και θέματα κοινωνικού αποκλεισμού. Κίνδυνο ένδυα σε ό,τι αφορά του πιο ηλικιωμένου πολιτές τη κοινωνία μας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δράσουμε πιο συστηματικά. Σκεφτόμενοι τώρα το μέλλον το μέλλον της ε, κοινωνικής πολιτικής και τη σύνδεση με το θέμα για το ζήτημα της ισότητας. Αυτό αποτελεί βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικό στόχο. Εδώ δεν χωράει αμφιβολία. Και δεν χωράει αμφιβολία το γεγονός ότι το gender mainstreaming, η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα. Και σκοπεύουμε στην κρατική προεδρία να τα προωθήσουμε. Εδώ θα πρέπει να δούμε μια πιο υγιή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα μέτρα και μέσα και θα χρειαστεί και μια συστηματική συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ όλων των δομών στην αρχή λοιπόν αυτού του θεσμικού κύκλου η πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήδη αναφέρθηκε, είναι σαφώς ένα θετικό σημάδι, μια θετική ένδειξη. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι έχουμε στοιχεία από διάφορες μελέτες και έρευνες αναφορικά με την ε, ισότητα των φύλων και θα πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες και οι μελέτες αυτές χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τα βαθύτερα αίτια των ανισοτήτων του επαγγελματικού και οικονομικού βίου, του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας και μια σειράς ολόκληρης προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά επίσης τη βία κατά των γυναικών γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα αυτό Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πρόκληση της ψηφιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης. Προστασία του κλίματος, παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη. Γι' αυτό λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στις εργασίες μας. Αν θέλουμε λοιπόν να επιμείνουμε στο σκέλος της βιωσιμότητας, το οποίο προφανώς έχει εκφραστεί ως στόχος, χρειαζόμαστε λοιπόν μια στρατηγική συστηματική προσέγγιση για όλες τις προκλήσεις αυτές. Να μην ξεχνάμε, ναι, ότι χρειάζεται μια ανεξάρτητη στρατηγική για την ισότητα. όπου και πάλι σκοπός ε, είναι η ενίσχυση της ε, ισότητας των φύλων και να επανέλθουμε στη σημασία της, ε, του κοινωνικού πλώνα, του πλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Και οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να συνεχίσουμε να ασκούμε την πολιτική ισότητα. Μία άλλη ερώτηση ακούσαμε. Αναφορικά με την αγορά εργασία. Εδώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. σα ευχαριστώ που το θέσατε ως ερώτηση. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και τα εμπόδια που εμποδίζουν τι γυναίκε για την συμμετοχή στην αγορά εργασίας. το θέμα της ε, φροντίδας μελών οικογενείας, το οποίο συνήθως επιφορτίζει τις γυναίκες. Αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο καλούμαστε να σκεφτούμε, να οργανώσουμε διάφορες πρωτοβουλίες. Και αυτό γιατί οι γυναίκες συχνά εργάζονται σε πιο μισθούς τομείς και σε πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί θα οδηγούσε σε, καλύτερη, σε καλύτερες συνθήκες και πιο πολύ ισότητα και σε πιο περιορισμένο κοινωνικό αποκλεισμό. Στα πλαίσια της ε, Κρατική προεδρία. προφανώ θα ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. και προς την κατεύθυνση αυτή θα διοργανωθούν διάφορες εκδηλώσει, το είπα αυτό και εισαγωγικά. Κάτι άλλο. Οι γυναίκες δυστυχώς δεν είναι σε πιο μειονεκτική θέση σε ό,τι αφορά του μισθού, αλλά και τι συντάξει Δυστυχώ αυτό αποτελεί μία επιπλέον πρόκληση. Το μισθολογικό και το συνταξιβετικό καθεστώς. Πόσο στα φτώχεια. Και αυτό προφανώ οδηγεί τι ε, γυναίκε σε μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη κοινωνικό αποκλεισμό. Επίλυση τέτοιων πολυσύμφετων φαινομένων και ζητημάτων ε, προαπαιτεί την συμμετοχή και τη δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων προφανώς ε, θα πρέπει με συνέπεια να εφαρμόζονται όλες οι διτάξει τη νομοθεσία από την πλευρά αυτή. Αναμένουμε και προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια για τις μισθολογικέ αποδοχές και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις για την ισότητα των δύο φύλων. Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά την διάσκεψη της ε, Κωνσταντινούπολης. Ακούσαμε μια ερώτηση. Η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί τμήμα του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αγωνιστεί για την πάταξη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Και 28 χώρες λοιπόν προσυπέγραψαν την ε, διακήρυξη αυτή. 21 μέλη την έχουν επικυρώσει και τα ε, προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή με την γνωμοδότηση της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2020. Καταρχάς, αναμένονται τα αποτελέσματα. Θα γίνει μια παρουσίαση για την υλοποίηση της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης. Θα συνεργαστούμε και με το Ινστιτούτο ισότητα σε ό,τι αφορά την βία καρτογενικών και στα πλαίσια της Προεδρίας θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου η επικύρωση του σημαντικού αυτού εγγράφου να ολοκληρωθεί, να είναι πλήρης, προκειμένου να καταστεί τμήμα της νομοθεσίας μας. Όπως σας είπα, αναμένουμε γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όμως πρώτα. Είμαι πεπισμένη ότι και η επόμενη Προεδρία θα επιμείνει στην υλοποίηση των ζητημάτων αυτών. Ευχαριστούμε πολύ για τι αναλυτικέ απαντήσει. Έχουμε δεύτερο γύρο. Η Λίνα νιώθω απευθεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις. Έχω δύο ερωτήσεις, μία πολύ σύντομη και μία λίγο πιο ε, εκτεταμένη ο πρόγραμμά σας λέτε ότι η ε, Κροατική Προεδρία θέλει να έχει ένα πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο φιλόδοξο. Θα ήθελα να ξέρω πώς μεταφράζεται αυτή η φιλοδοξία ε, όσον αφορά τις πολιτικές ισότητε. Και η δεύτερη ερώτηση είναι διότι εσείς τονίσατε κυρίως ότι θα πρέπει να εντάξουμε τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δημογραφικά προβλήματα. Αλλά ε, αν επικεντρωθούμε μόνο ε, στα όσα έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας, δεν θα λύσουμε τα δημογραφικά προβλήματα και ούτε θα λύσουμε και τα προβλήματα ισότητας, διότι εκτός και αν προσπαθήσουμε ταυτόχρονα να δούμε ε, και κατάλληλο καταμερισμό χρόνου εργασίας και αφοσίωση στην οικογένεια, οι άντρε και οι γυναίκε δεν θα μπορούν να ενταχθούν ισότιμα στην αγορά εργασία, γιατί ενταχθώ, εντασσόμαστε με τελείω διαφοροποιημένο τρόπο και ιδίω διαφοροποιημένο μεταξύ των γυναικών, ανάλογα με το εισόδημα, ε, από το που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλαίσιο κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουμε να έχουμε καλύτερο καταμερισμό χρόνου εργασίας και οικογενειακής ε, ζωής. Εδώ δεν βλέπω τίποτα στην πρόταση, για παράδειγμα, όσον αφορά την προώθηση ε, ισότιμων αδειών που δεν είναι μεταβιβάσιμες και αποζημιώνονται στο 100% μεταξύ ανδρών και γυναικών, πατέρα και μητέρας δηλαδή. Δηλαδή, να μην μπορούν να μεταβιβάσουμε την ε, άδεια πατρότητας και μητρότητας. Επίσης, όσον αφορά την ε, προαγωγή των δημόσιων υπηρεσιών, αναφέρεστε ε, στα όσα ε, θα πρέπει να προσέχουμε στη διάρκεια της ζωής μας για την υγεία, αλλά έχουμε και πολλά πράγματα ε, τα οποία αφορούν την παιδική ηλικία. Επίσης, πιο ισότιμη εκπαίδευση. Τα όσα είπε η συνάδελφος η Μαρία Οχένια Παλόπ για κάποιες αξίες οι οποίες δεν είναι και ακριβώς ισότιμες αν θα προωθήσετε και συγκεκριμένα προγράμματα για να ενταχθούν περισσότερο οι γυναίκες ε, στις ε, τεχνολογίες για μια ψηφιακή επανάσταση όπου οι καλύτερα αμοιβόμενε εργασίες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε άντρες ε, και αυξάνεται το μισθολογικό χάσμα. Και τέλος, εσείς αναφερθήκατε επίσης και στη συνέργεια μεταξύ κοινωνικών πολιτικών και οικονομικών πολιτικών. Θα ακολουθήσει η Κροατική Προεδρία τη στήριξη στις ε, οικονομικές πολιτικές ε, ε, περικοπών λόγω πληθωρισμού. Δεν ευνοούν σε καμία περίπτωση ε, τις υπηρεσίες. μειώνουν τις υπηρεσίες φροντίδες, όπου είμαστε οι βασικές οι οποίες παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες και επομένω είναι πάρα πολύ αρνητικός ο αντίκτυπος για μας. Ευχαριστώ. Η η Μπελίντα Ντελούση. Καλωσορίσατε κυρία Υπουργή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να καταμαλωμήσετε αυτό το οποίο θα αποκαλούσα εγώ ε, φεμινισμό υπό όρους ε, και ε, επιλεκτική προσέγγιση που πλήττει τις γυναίκες αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, οι ομάδες ε, φεμινιστριών δεν μιλάνε... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Μισό λεπτό να το ελέγξουμε. Could you please repeat? μπορείτε να τα ξαναπείτε. Ναι, ναι, ωραία, θα ξαναρχίσω. Ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα και το χρόνο που μας αφιερώνετε. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να καταπολεμήσετε αυτές τις οποίες αποκαλώ ε, φεμινισμό υπό ε, και επιλογή ε, οργή, η οποία πλήττει τα, τις ομάδες γυναικών. Για παράδειγμα, οι φεμινίστριες δεν μιλούν για τις χιλιάδες μικρές κοπέλες οι οποίες βιάζονται ε, και βασανίζονται από ε, πατριαρχικούς πολιτισμούς που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πολιτιστικό το πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν λένε τίποτα και μάλιστα ένας εργατικός ε, βουλευτής που μίλησε χρειάστηκε να παραιτηθεί και έχασε και τη θέση της. Και η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουμε περιπτώσεις, για παράδειγμα, ε, όπου φεμινίστρες μιλάνε, ε, για παράδειγμα, το δικαίωμα των γυναικών να φοράνε το χιτζάμπ άμα θέλουν, αλλά δεν λένε ότι οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να το φορούν και ορισμένες φορές μπορεί και να τις φυλακίσουν, να τις βασανίσουν, να τις βιάσουν εάν δεν το κάνουν. Φαίνεται να οργιζόμαστε για κάποια σχόλια που μπορεί να έκανε ο Τραμπ επειδή ε, θόπευσε μια γυναίκα, ε, ενώ δεν έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για άλλα θέματα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά σε πολιτιστικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια και να μην επιλέγουμε να υποστηρίζουμε κάποια προβλήματα απλώ και μόνο οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες νιώθουμε ότι μπορούμε να θίξουμε κάποια θέματα. Αυτό είναι έλλειψη τόλμης και απογοητεύουμε πολλές γυναίκες και νέες κοπέλες. Ε, πρέπει να ε, έχουμε το θάρρος να λέμε την αλήθεια και πραγματικά θα ήθελα να ξέρω και ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτό τον επιλεκτικό φεμινισμό, ο οποίος φαίνεται να προστατεύει κάποιους άντρες από οποιαδήποτε δίωξη και αφήνει τις νέες κοπέλες ε, έρμεο σε οποιαδήποτε ε, συμπεριφορά. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ Κάποιες σύντομες ε, ερωτήσεις. Οι συνέπειες ε, της ε, κλιματικής επιλής αφορούν κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά. Πρόσφατα στο Κοινοβουλίο συζητήσαμε το θέμα της Πράσινης Συμφωνίας. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπό την Κροατική Προεδρία, εσείς θα είστε μια ισχυρή φωνή που θα λάβει υπόψη την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Και ενώ θα οικοδομείτε τις πολιτικές, θα λάβετε υπόψη και θα μιλήσετε ε, ισχυρά εκ μέρους των γυναικών για να χρησιμοποιηθεί και η εμπειρία των γυναικών. Έχετε πει πολλά για την προστασία των αναπαραγωγικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων των γυναικών και για την κοινωνική πολιτική. Όμως νομίζω ιδιαίτερα σχετικό εδώ είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι σημαντική και η εκπαίδευση εδώ και η σεξουαλική εκπαίδευση είναι μορφή παιδείας. Γιατί λέγονται όλο ένα και λιγότερα για τα φροντίσια νοσήματα, το AIDS, τις πρώιμες εγκυμοσύνες ε, και τα λοιπά και η βοήθεια προς τις γυναίκες δεν μεταφράζεται πάντοτε προς τη στήριξη του οικονομικού τους καθεστώτος. Οι γυναίκες, παραδείγματος χάρη στην Πολωνία, λαμβάνουν χρήματα ε, ως ε, υποστήριξη των παιδιών και ε, ως αποτέλεσμα αυτού 100.000 γυναίκες ε, εγκατέλειψαν την εργασία τους Φανταστείτε λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιε είναι οι συνέπειες για τις ε, συντάξεις των γυναικών αυτών ή όταν θα θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, τι προβλήματα θα έχουν. Επομένως, ε, κάθε κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι ισορροπημένη και καλά σχεδιασμένη και θα πρέπει να βοηθά τις γυναίκες να επανέρχονται στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Γιατί Ποιο είναι το ενδιαφέρον, παραδείγματο χάρη, η Κροατία έχει ένα καλό σύστημα αρρωγή ε, των νέων μητέρων. Βλέπετε από τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος, παραδείγματο χάρη, οι γυναίκες να κάνουν παιδιά πριν τα 40 έτη τους και είναι χρήσιμο για να μπορέσουν οι γυναίκες να επανέλθουν στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Thank you very much and finally... Ευχαριστώ και τέλος θα θέσω και εγώ μια ερώτηση. Και πάλι θα αναφερθώ στο θέμα της συμβατότητας, της επαγγελματικής και ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχουν ε, οικονομικές εγκαταστάσεις μέρημνας και αυτό είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ε, και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το χάσμα στις ε, συντάξεις, το μισθολογικό χάσμα και θα πρέπει να προωθήσουμε τη γεννητικότητα. Να δούμε τις στατιστικές. Ε, οι χώρες όπου οι γυναίκες μπορούν να πούνε ότι θέλω μία ασφαλή δουλειά και απασχόληση είναι εφικτό εάν ε, μπορούν να προσαρμόσουν και το χρόνο εργασία τους. Ε, δηλαδή αυτό έχει να κάνει με αυτά που είπε η Ελιζαμπέτα. Με ενδιαφέρουν ε, όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και τα εργαλεία που προτείνετε εσείς. Μπορείτε να αναμένετε μία αναβίωση των στόχων της Βαρκελόνης. Με ενδιαφέρει να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε εκεί. Υπήρξε και μια αναφορά στα συμπέρασμα του Συμβουλίου. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν πραγματικέ υποχρεώσει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Με ενδιαφέρουν λοιπόν τα εργαλεία, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε σε αυτό το έργο. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά τις γυναίκες και τους άντρες στα διοικητικά συμβούλια. Θα υπάρξει κάποια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ που θα απαντήσετε τις ερωτήσεις μας. Μάλιστα, να κάνουμε πάλι μια ομαδοποίηση των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Είναι σημαντικά τα ζητήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ισότητας, την ισότητα των γυναικών, στην αγορά εργασίας. Και να ξεκινήσω από τις τελευταίες ερωτήσεις. Να απαντήσω λοιπόν πρώτα στη δική σας ερώτηση, κυρία Πρέτρε. Οι γυναίκες ε, στα συμβούλια. Ξέρουμε ότι ο φάκελος αυτός έχει μπλοκαριστεί. Τα επόμενα δύο χρόνια στο Συμβούλιο ε, δεν έγιναν διάφορες συζητήσεις. Το κείμενο είναι έτοιμο βέβαια, αλλά όπως έχουν τα πράγματα δεν έχουμε κάποιο λόγο να πιστεύουμε ότι ότι θα αλλάξουν τη γνώμη, α, ε, τη γνώμη τους οι χώρες που μπλοκάρουν το, το ζήτημα αυτό αν ε, υπάρξει κάποιο κάποια αλλαγή, προφανώς και θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε το ρόλο μας για να πετύχουμε μια μεγαλύτερη τεκρότητα και πιο σωστή αντιμετώπιση. Το ερώτημα για το πι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το θέμα αυτό αποτελεί, αν θέλετε, και το πλαίσιο για πολλές άλλες ερωτήσεις που ακούσαμε. Και φυσικά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από πολιτικής άποψης είναι το πιο σημαντικό θέμα. Το πιο σημαντικό ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους, ή η Κρατική Προεδρία τους επόμενους ε, μήνες. Και ελπίζουμε λοιπόν να βρούμε ένα συμβιβασμό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ελπίζουμε να βρούμε λοιπόν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τοποθέτησης ε, των συντηρητικών δυνάμεων που επιθυμούν πιο πολλά δημοσιονομικά μέσα. Μάλλον εκείνων που χρειάζονται πιο πολλά δημοσιονομικά μέσα και εκείνων που θέλουν να υπάρχουν πιο λίγε δαπάνε στο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά λαμβάνοντα υπόψη την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμεί λοιπόν ε, είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε υπόψη όλε αυτέ τι ανησυχίε αλλά και όλε τι ανάγκε των κρατών μελών. Βασιζόμαστε λοιπόν στην κοινή συνεργασία και στο υψηλό επίπεδο δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Θα πρέπει προφανώ ε, να μείνουμε όσο πιο ουδέτεροι γίνεται και προ την κατεύθυνση αυτή η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και στους κόλπους του Συμβουλίου στην εξέβρεση συμβιβασμών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και ασφαλώς. Να επαναλάβω ότι θα χρειαστεί ένα συμβασμός που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υλοποίηση ενός προγράμματος φιλόδοξου. Και θα θέλαμε να συνεχίσουμε φυσικά να χρηματοδοτούνται όλες οι πολιτικές που κατοχυρώνονται στις ε, συνθήκες, η πολιτική για την ε, γεωργική ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή και φυσικά να λάβουμε υπόψη όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τηρήσουμε λοιπόν την ενότητά μα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι διαφορέ που υπάρχουν, πολιτισμικέ δημογραφικέ και ούτω καθεξή. Ο συμβιβασμό λοιπόν αυτό θα πρέπει να λειτουργεί ε, σωστά για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Επαναλαμβάνω όμω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν σε κάθε χώρα διαφορετικές ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχέση, τη σχέση μεταξύ του ΠΔΠ και το θέμα του κράτους δικαίου, το θέμα αυτό είναι βασικό και θεμελιωδού σημασία. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις σε ό,τι αφορά την, τα εμπόδια που έχουν οι γυναίκε για πρόσβαση στην αγορά εργασία. Και το γεγονό ότι έχουμε ότι συχνά δεσμεύονται να φροντίζουν για τα μέλη τη οικογένεια. Και το γεγονό ότι συχνά θεωρείται ότι δεν είναι εξίσου ικανέ για τη δουλειά όπω οι άντρε. Και η λύση για τέτοια προβλήματα προφανώς θα συνέβαλε και στην μεγαλύτερη ισότητα των δύο φύλων και έτσι αυτό με τη σειρά του θα μείωνε τον κοινωνικό αποκλεισμό και την πιο υψηλή προφανώς θα οδηγούσε σε πιο υψηλή οικονομική ανάπτυξη. Μιλώντας για την κρατική προεδρία, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες ανέφερα και εισαγωγικά για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, λοιπόν. Τα πολύ αυτά ζητήματα προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συστηματικό τρόπο. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω εκ νέου ότι θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι φορείς θα πρέπει να εκτελεστούν και να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας και αναμένουμε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα τη στρατηγική ισότητα και για την διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι μισθολογικέ αποδοχέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ισότητα γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασία και το θέμα των μισθολογικών αποδοχών, μίλησα για το θέμα των συντάξεων, το οποίο ε, αποτελεί εξίσου μεγάλο ζήτημα. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο διαφορά σε ό,τι αφορά τους μισθούς, αλλά και τις συντάξεις. Οι συντάξεις λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστούν με καλύτερο τρόπο να αποτελούν, να είναι πιο βιώσιμες και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο προφανώς τα συστήματα συνταξιευότησης προφανώς και αποτελούν ε, εθνική αρμοδιότητα. Αλλά είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε μια σωστή σύνταξη και προφανώς ε, και οι γυναίκες και οι άντρες έχουν ίση, ίσα δικαιώματα προκειμένου να έχουν σωστά εισοδήματα στην μεγαλύτερες ηλικίε προκειμένου να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη φροντίδα των μελών της οικογένειας και το θέμα της, ε, του συνδυασμού της φροντίδας αυτής με ένα επάγγελμα. Θα αναμένουμε και τις, ε, τα πορίσματα του Συμβουλίου για το πώς μπορούν αυτοί τα στοιχεία να συνεπάρξουν. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προωθήσουμε το σκέλος αυτό στην οικογένεια, τη ε, συμμετοχή των γυναικών. γιατί το σκέλο τη φροντίδα των μελών οικογένεια είναι ένα καταλητικό παράγοντα για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Και θα πρέπει γενικά ο Ευρωπαίο πολίτη να είναι πιο καλά ενημερωμένο για τα εφιστάμενα μέτρα. Τα οποία βοηθούν ακριβώ στην συμφελίωση επαγγελματικού και οικονομικού και οικογενειακού βίου. Και θα βασιστούμε στα πορίσματα του Συμβουλίου και σε ένα έγγραφο, σε μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητα και θα συμμετέχουν ε, φυσικά και όλοι οι φορείς που θα συμμετέχουν στη διάσκεψη για τα δικαιώματα των γυναικών. Ένα άλλο ερώτημα. Ποιοι είναι οι στόχοι της Βαρκελόνης. πρόεδρος ε, επισημαίνει ότι δυστυχώς δεν έχουμε πολύ ώρα ακόμα μπροστά μας. Αν ναι, σωστά κατάλαβα, πρέπει να ολοκληρώνω. Έχουμε μόλις λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Η ε, στόχη της Βαρκελόνης, λοιπόν, όπως ε, αναφέρθηκε. θα τους επιδιώξει στην ε, Προεδρία, τη ε, Κρατική Προεδρία, σε ό,τι αφορά και το θέμα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει προφανώς σε όλα τα επίπεδα να αναλάβουμε δράσεις. για να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών. Υπάρχουν και άλλες μορφές βίας, δυστυχώς σεξουαλική βία. Εξαιρετικά επιβλαβείς πρακτικές. Έχουμε επίσης και ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες γυναικών. Να μην ξεχνάμε και τις γυναίκες με αναπηρία στο πλαίσιο αυτό. Δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε για την ομάδα αυτή. αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα και συχνά είναι θύματα βίας. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και τις ε, πληροφορίες, τα στοιχεία που μας έδωσε η κυρία Ντάλη σε ό,τι αφορά τη νέα στρατηγική για την ισότητα των φίλων. Το Μάρτιο. Και θα υπάρξουν εκδηλώσεις και μέσα και μέτρα για την καλύτερη προστασία των γυναικών και την μεγαλύτερη ισότητα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τις γυναίκες και τα παιδιά. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να συνεχίσω. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ήταν όλες εξαιρετικά σημαντικές. Και ασφαλώς ε, να είστε σίγουροι ότι η κρατική προεδρία θα προωθήσει όλα τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ. Σίγουρα έχουμε μία ευρεία εικόνα σχετικά με όλα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ολοκληρώνουμε εδώ. Θα διαβάσω όμως τις ανακοινώσεις για το πρωτόκολλο. Όλο αποφασίσαμε κατά τη συναντρίαση των συντονιστών στις 4 Δεκεμβρίου 2019 θα σταλούν έτσι ώστε θα τα έχετε γραπτός γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό αποφάσεων σε σχέση με τις γνωμοδοτήσεις και τι πρέπει να κάνουμε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστούμε πολύ την προσκεκλημένη μας. Σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στην Προεδρία σας και φυσικά μια καρποφόρο συνεργασία μεταξύ Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και με όλα τα θεσμικά όργανα. Καλή επιστροφή και καλή δουλειά για το απόγευμα.